εγκασμένη να αποτύχει, ποτέ δεν πρόκειται να περάσει και η μόνη σωστή πολιτική λύση είναι να την αποσύρουμε. Ευχαριστώ. Ε, Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Μετά τη συζήτηση ε, κατατέθηκαν τέσσερις προτάσεις ε, ψηφίσματος. Έκλεισε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε σήμερα το θέμα αυτό στις 12 η ώρα. Προχωρούμε στη μερίσια διάταξη στο σημείο που αφορά την κατάσταση των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Είναι μια προφορική ερώτηση και δίνω το λόγο στο συντάκτη, στον κύριο Μορέιρα, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για μια προφορική ερώτηση που την ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και ως πρόεδρος εγώ είμαι ε, το φερέφωνο της Επιτροπής και παρουσιάζω την προφορική ερώτηση της ΣΥΝΤΑ. Οι διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ επανελήφθησαν επίσημα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ το 2010 μετά από πολλά έτη διακοπής. Ο στόχος είναι να ε, επιτευχθεί διαπραγμάτευση για μια συνολική εμπορική συμφωνία. Εννέα γύρι διαπραγματεύσεων έχουν λάβει χώρα έκτοτε. Μέχρι σήμερα, εν λόγω γύρι έχουν επικεντρωθεί στο κανονιστικό τμήμα τη συμφωνία, Ενώ δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία για την ανταλλαγή των προσφορών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Γιατί ε, χωρί το σημείο αυτό δεν υπάρχει ουσιαστική διαπραγμάτευση. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει μια λεπτομερή εικόνα τη κατάσταση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μερκοσούρ. Μια και έχουν περάσει πάνω από δύο έτη από την επίσημη επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνία σύνδεση. Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν επί το παρόντο οι διαπραγματεύσει. Πού προσκρούν. Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει του βασικού στόχου και να αναφέρει ποιε είναι οι προσδοκίε για την επόμενη Υπουργική Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του Ιανουαρίου 2013 και θα γίνει στο Σαντιάγο τη Χιλής. Αυτό είναι το κείμενο της προφορικής ερώτησης Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου. Θα ήθελα τώρα Ω πρόεδρο τη Επιτροπή, να επιβάλλω και μερικέ παρατηρήσει επιπλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικό εμπορικό εταίρο του Μερκοσουρ, 20% του συνολικού εμπορίου με το Μερκοσουρ και είναι και ο πρώτο επενδυτή στην περιοχή. Ε, είναι σημαντικές οι άμεσες ε, αλλοδαπές επενδύσεις, πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα το Μαρκοσούρ είναι 8ος ε, εμπορικό εταίρο Ένωση. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση των εμπορικών σχέσεων από 28 δίστα το 2007 στα 45 δισεκατομμύρια τζίρο των εμπορικών διαπραγματεύσεων το 2008. Σημαντική λοιπόν σε τι αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την περιοχή του Μερκοσούρ. Είναι ε, σκόπιμη λοιπόν η σύναψη εμπορική συμφωνία με την περιοχή του Μερκοσούρ, γιατί είναι σημαντικό το δυναμικό ανάπτυξη αυτών των εμπορικών σχέσεων, όπω φάνηκε και από την ανάπτυξη που σα παρουσίασε. Φαίνεται όμω ότι η είναι πολύ δυσίωνη η κατάσταση. εδώ καταραμένη αυτή η εμπορική συμφωνία. Ξεκίνησαν πριν από μία δεκαετία. Διακόπηκα στη συνέχεια θεωρώντα ότι δεν υπήρχαν πρόσφορε συνθήκε για την σύναψη συμφωνία. Ε, δόθηκε μία τόνωση από την Ισπανική Προεδρία. Πάλι έχουμε φτάσει σε διέξοδο. Υπάρχουν πολέμοι και από τις δύο πλευρές που μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, με τις ε, εξελίξεις στο Μερκοσούρα ε, τα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Τα μέτρα προστατευτισμού και η κατηγορηματική θέση κάποιων ε, χωρών της Λατινικής Αμερικής κατά της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δυστυχώς δεν, δυστυχώς δεν προϊονίζονται θετικές εξελίξεις για την εμπορική συμφωνία. Φαίνεται ότι το Μερκοσούρ θέλει να μετατραπεί σε μια εσωστρεφή οικονομία και δεν συμμετέχει στην τάση φιλελευθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου. Φαίνεται ότι στη Λατινική Αμερική υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, Κολομβία, Περού, Χιλή, Μεξικό έχουν εκδηλώσει ένα εμπορικό άνοιγμα και προθυμία σύναψη εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα όλε αυτέ οι χώρε έχουν διμερεί εμπορικέ συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στο Μερκοσούρ η Βραζιλία, Αργεντινή και άλλε χώρε έχουν βρεθεί εκτός ε, αυτής της προσπάθειας εμπορικού ανοίγματο. Και μάλιστα οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και η ακινητοποίηση των διαπραγματεύσεων, το, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ακριβώ αυτή τη διάσταση απόψεων που υπάρχει και δυστυχώ μία ζωφερή εξέλιξη και ζωφερέ προοπτικέ για το μέλλον. Η προφορική ερώτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει κάποιες ε, κρυμμένες ε, άδειλες ε, προθέσεις ή προτάσεις. Απλώς διαρωτόμαστε, έχει νόημα να συνεχίσουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις αν δεν υπάρχουν ελπίδες να διεκπεραιωθούν, να έρθουν σε αίσιο πέρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι για να τροποποιήσει τα δεδομένα και να πείσει τους τέρους του Μερκοσούρ ε, να τροποποιήσει τη θέση τους. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να ευοδοθούν τελικά αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά δυστυχώς ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητες να προχωρήσει την κατάσταση, αλλά είναι πραγματικά ένα σημαντικό εταίρο του Μερκοσούρ. Είναι προ το συμφέρον μα να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία και νομίζω ότι είναι και προ το συμφέρον του Μερκοσούρ. Θα πρέπει να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Σιγητά, το λόγο τώρα έχει ο Επίτροπο κ. Στεχόχτ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ δεν σήμεσαν την πρόοδο που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δουλέψαμε παρόλα αυτά από τη στιγμή που ξαναρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις το 2010. Και μάλιστα το ίδιο το Μερκοσούρ μας ζήτησε να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις οι, μέχρι στιγμής αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν εστιάσει στο καονιστικό τμήμα της συμφωνίας, δηλαδή στους βασικούς καόνες και στις αρχές που θα αποτελέσουν τη βάση για τις δεσμεύσεις των δύο πλευρών ε, και την δυνατότητα να ανοίξουν τις αγορές τους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολύτιμα κεφάλαια στους καόνες καταγωγής και στις ε, υπηρεσίες ε, και επενδύσεις στις υπηρεσίες αλλά δεν έχουμε μπει στην καρδιά του θέματος, δηλαδή στην πραγμα... στο πραγματικό θέμα της πρόσβασης της αγοράς του ενός στο... στην αγορά του άλλου. Στις ε, κρατικές προμήθειες και στις ε, επενδύσεις ε, στις υπηρεσίες για την κατάργηση των φραγμών. Αυτή η προσέγγιση έφτασε τα όρια της, όπως αναγνώρισαν και οι δύο πλευρές στο τέλος του τελευταίου διαπραγματευτικού γύρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο τώρα είναι μέσω ανταλλαγής προσφορών για πρόσβαση στην αγορά για τις ε, δημόσιες ε, προμήθειες, ε, τα αγαθά, τις υπηρεσίες. Αλλά το Μερκοσούρ δεν έχει συμφωνήσει στο εσωτερικό του για το πώς θα προσφέρει αυτή την πρόσβαση στην αγορά. την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μία συνάντηση με τους ομολόγους μας στο, στο Μερκοσούρ, στην, στο Σαντιάγκο της Χιλής, 26 Ιανουαρίου, σε μία σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θα είναι μία ανταλλαγή σε υψηλότερο επίπεδο. Οι διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ είναι περίπλοκες και αυτό έχει επιπτώσεις και στις διαπραγματεύσεις. Καταρχάς, ποια χώρα είναι μέσα και ποια είναι έξω από το Μερκοσούρ η Παραγουάη, η, μελλοντική διεύρυνση στη Βολιβία ε, μπορεί να περιπλέξει ε, σε κάποιο βαθμό τα πράγματα. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις στο εσωτερικό του Μερκοσούρ. Σε τμήμα του Μερκοσούρ υπάρχουν ε, αυξανόμενες τάσεις για υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού, που μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορούν πραγματικά να έχουν ανοιχτή αγορά. Στην επόμενη υπουργική συνάντηση στο Σαντιάγκο της Χιλής θα καταγράψουμε την κατάσταση και θα έρθουμε σε επαφή με τους ε, ομολόγους μας, ούτως ώστε να συμφωνήσουμε για το τι χρειάζεται, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, παρά τις δυσκολίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη για τις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να υπάρξει μια ισορροπημένη και φιλόδοξη συμφωνία ε, με το Μερκοσούρ. Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να έχει ωφέλη και για τις δύο περιοχές. Σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις. Να είστε σίγουροι. Ετοιμάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής στο Σαντιάγκο, Συζήτησα το θέμα με τους συναδέλφους ε, στην περιοχή. Και η αίσθησή μας είναι ότι έχουν δυσκολίες να καταλήξουν σε προτάσεις προσφορών για το άνοιγμα των αγορών. Δεν θα είναι έτοιμοι μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο. Παρόλα αυτά, δεν θέλουν να σταματήσουν διαπραγματεύσει, γιατί ξέρουν ποιε θα ήταν οι πολιτικέ συνέπειε αυτού. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αποφασίσουν ή θα κάνουν διαπραγματεύσει για ελεύθερο εμπόριο και δεν θα είναι εύκολο για αυτού, αλλά ούτε και για εμά να προτείνουμε κάποιε προσφορέ για άνοιγμα αγορών. Ή α, θα ξεχάσουν τη συμφωνία. Και τα δύο δεν γίνονται. Ε, θα πρέπει και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση του επόμενου μήνε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ή θα κάνουμε, θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε ενώπιον του ΠΟΕ για το θέμα αυτό. Είναι σαφές ότι για διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί, για διάφορους κανονισμούς που έχουν προχωρήσει, στους οποίους έχουν προχωρήσει κάποια κράτη-μέλη του Μερκοσούρ, όπως η Αργεντινή, αλλά όχι μόνο η Αργεντινή, έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή, ας πούμε για τις υπηρεσίες. θα πρέπει κάποια στιγμή να επιχειρηματολογήσουμε λογικά και να σημειώσουμε πρόοδο. Όταν γίνει η συνάντηση που σας προανήγγειλα θα σας ενημερώσω για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Σαλαφράγκα πρώτος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι είναι πολύ ε, σκόπιμη η συμπερίληψη αυτής της συζήτηση σήμερα εν ώψη της ε, διάσκεψης κορυφής ε, της ΕΛΑΚ στο Σαντιάγο της Χιλής την επόμενη εβδομάδα. Με τη Χιλή έχουμε εμπορία σύνδεσης με καταπληκτικά αποτελέσματα. Το Δεκέμβριο κυρώσαμε την πολυμερή συμφωνία με την Κεντρική Αμερική. Ακόμη και με την Κούβα έχουμε εξελίξεις θετικές. Και μάλιστα εν ώψη της διάσκεψη κορυφή Μαδρίτη, ε, εγώ συζητητή ε, τη Συμφωνία Σύνδεση, ε, επισκέφθηκα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μίλησα με τον κύριο Ντεχούχτ, με τον Επίτροπο, προκειμένου να ξεμπλέξουμε τι διαπραγματεύσει. Είναι δεδομένο το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ μια ισορροπημένη και φιλόδοξη συμφωνία, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι ευαισθησίε και τα λεπτά σημεία του θέματο. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε στην πολιτική κατάσταση στο Μερκοσούρ. Όντως, μετά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων και εξαιτίας του Μερκοσούρ δεν καταφέραμε να θέσουμε επιτάπητος μια προσφορά που να βελτιώνει τη διαπραγματευτική προσφορά του 2008. Γνωρίζουμε την κρίση στην Παραγουάη, ε, την συμπερίληψη της Βενεζουέλας, ε, την αναστολή ως προς την Παραγουάη και γνωρίζουμε ότι το θέμα των ευαίσθητων προϊόντων αφορά το 10% μόνο των εμπορικών συναλλαγών. Κύριε Επίτροπε, θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους των χωρών του Μερκοσούρ για τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας. Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα, όπως επισημάνατε, ότι δεν υπάρχει τέτοια πολιτική βούληση, ποιες θα ήταν οι εναλλακτικέ λύσεις. Θεωρείτε κύριε Επίτροπε ότι θα ήταν ευκταίο να συνάψουμε συμφωνία με εκείνες μόνο τις χώρες που εκδήλωσαν την ε, διάθεσή τους και την προθυμία τους να καταθέσουν ε, μια λογική διαπραγματευτική προ... πρόταση επιτάπητος, δηλαδή Βραζιλία, Ουρουάη, Παραγουάη. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει βούληση όλα είναι εύκολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σούστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως Επιτροπή ΙΝΤΑ θελήσαμε να προκαλέσουμε μία συζήτηση στο Κοινοβούλιο γιατί μας φαίνεται σημαντικό εν ώψη της Συνόδου Κορυφής μεταξύ των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινική Αμερική και εν ώψη της Eurolat που θα ξεκινήσει ε, στο Σαντιάγκο τη Χιλή σε λίγε μέρε, είναι σωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μια κατεύθυνση ε, και να δώσει και την άποψή του για αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο θέμα εμπορικών ανταλλαγών. Η σχέση μεταξύ Ευρώπη και αυτού του τμήματο Λατινική Αμερική εντάσσεται στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ατλαντικών δυνάμεων. Σε μια εποχή μεγάλου ανταγωνισμού, σε μια εποχή μεγάλης παγκοσμιοποίησης, η Ευρώπη έχει ανάγκη από στρατηγικές συμμαχίες. Μην ξεχνάτε την συμφωνία με το Μεξικό, τη Χιλή, το Περού. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματικό συμφέρον να ξεκινήσει σημαντικές πρωτοβουλίες απέναντι σε αυτή την περιοχή του πλανήτη για να δημιουργήσει μια μεγάλη περιοχή ανταλλαγής εμπορικών αγαθών. Ξέρουμε πολύ καλά τα, τους φραγμούς, καταλαβαίνω τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρω ότι ενημερώσατε και το Κοινοβούλιο Νομίζω όμω ότι πρέπει να είμαστε πολύ σταθεροί και να δείξουμε ποια είναι τα όρια, ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, τι έκανε τα τελευταία χρόνια η Αργεντινή και άλλε χώρε Να μην ξεχνάμε τι προστατευτικέ τάσει και τη Βραζιλία, που είναι εμπόδιο στην επανέναξη αυτή τη στρατηγική, που είναι όχι μόνο εμπορική αλλά και πολιτική. Ούτως ή άλλως Ούτω η άλλω το εμποριο ειναι μια ειναι η αιχμη του δόρατος μια πολιτική στρατηγική. Θέλουμε να δώσουμε λοιπόν ως ένα σήμα, ένα μήνυμα ως Κοινοβούλιο ε, ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και μπορούν να φτάσουν σε μια πραγματική ανταλλαγή προσφορών για το άνοιγμα των αγορών. Ευχαριστώ κύριος Μετίν Καζάκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη λύπη μας για την έλλειψη ουσιαστικής προόδου στην υπόθεση των συναλλαγών Μερκοσούρ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από πλευράς των πολιτικών. Ορισμένα κράτη έχουν προβεί σε συνεννοήσεις και ρυθμίσεις ε, σε περιορισμούς των προμηθειών, ε, ε, περιορισμούς στην επιβολή φόρων σε εξαγωγές η μη ε, αυτόματη αδειοδότηση κοστίζει 45 εκατομμύρια ευρώ στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει επανακρατικοποιήσει ε, την ενέργεια και ε, έτσι καταπατά τις δεσμεύσεις της πολέμηση του προστατευτισμού και στέλνει και αρνητικά μηνύματα στους ξένους επενδυτές. Πέρα από αυτά τα αρνητικά σημεία όμως, θα πρέπει να τονίσουμε και κάποια θετικά. Οι δύο περιφέρειες δεσμεύονται να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συμφωνία αυτή θα σημάνει 4,5 δις ε, ε, όφελος και για τις δύο πλευρές. Εμείς οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, οι δημοκρατικοί κανόνες, η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι ένα απόσπαστο τμήμα τη συμφωνίας αυτής. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ολοκληρωμένη πολιτική και να υπερασπίζεται τα οικονομικά της συμφέροντα, αλλά και να προωθεί τις δημοκρατικές της άξιες, θα πρέπει να είναι πιο στεναρή στι τάσει κατά τη διάρκεια τη επικειμένη Συνόδου Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμέρική. Συμπέρασμα. Ε, θέλουμε μία προσέγγιση με μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο δομημένη για να καταπολεμήσουμε τα εμπόδια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέζ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και μία δεκαετία έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ. Και όπως και με τις συμφωνίε για την Κολομβία, το Περού, την Κεντρική Αμερική, έχουμε τις ίδιες φιλελεύθερες ε, συνταγέ επιτάπητο. Ε, δηλαδή, ε, μια τρομερή ανισορροπία μεταξύ των δύο περιοχών. εισαγωγή τρίτων πρώτων υλών και γεωργικών προϊόντων, που ουσιαστικά ε, ε, σαρκώνουν το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως συντοβολώνα της Ευρώπης εις βάρος ε, των γεωργών και των δύο πλευρών. Και απ' την άλλη εξαγωγή πρώτων υλών και υπηρεσιών. Ούτε και εκεί έχουμε τις αναμενόμενες και επιθυμητέ εξέλιξεις. Μας προτείνεται τώρα ένα ψήφισμα για να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις με τον Μαρκοσούρ εν ώψη της διάσκεψης που που θα λάβει χώρα στα τέλη του μηνός. Η πολιτική ομάδα είναι κατά του ψηφίσματος. Δεν μας έχει διαφύγει ότι από το 1999 είχαμε σοβαρότατες πολιτικές εξέλιξεις στην περιοχή. Η Παραγουάη μετά το πραξικόπημα πολύ σωστά έχει, ε, ε, ε, έχει ανασταλεί η συμμετοχή της στο Μερκοσούρ. Βολιβία, Χίλια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εκουαδόρ, Περού. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση και αποτελματωμένες διαπραγματεύσεις αφενός και αφετέρου ρηξικέλευθες πολιτικές εξελίξεις. Ως η συγγήτρια της έκθεσης για τη βιοπειρατεία που εγκρίναμε στην αρχή της εβδομάδας, ε, ε, διαπιστώνουμε σημαντικό νομοθετικό ενδιαφέρον χώρες αυτές. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, για την πνευματική ιδιοκτησία που δίνει προτεραιότητα στο ελεύθερο λογισμικό και στα γενώσιμα. Δυστυχώς οι γεωγραφικές ενισορροπίες εξελίσσονται ραγδαία. Είναι αντιπαραγωγικές αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Ε, με... Είμαστε υπέρ των ισορροπημένων διαπραγματεύσεων και η λύση είναι απλούστατη και προφανή ε, να ξεκινήσουμε εξ αρχής διαπραγματεύσεις με τους σωστούς συνομιλητές. Ευχαριστώ κυρία Μακλάρκιν. Τα πιθανά ωφέλη μεταξύ μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοζού είναι τεράστια. Ε, μια συνδυασμένη αγορά πάνω από 800 εκατομμύρια καταναλωτών. Ε, Πάντω δεν έχουμε εξελίξει μετά από τρία χρόνια από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτική υποστήριξη και από τι δύο πλευρέ, ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει και οι δύο πλευρέ να είναι έτοιμε να ανοίξουν τι ε, αγορέ του με αμοιβαία υποφελή τρόπο. Ε, τα προστατευτικά μέτρα που παίρνουν κάποιες χώρες Μερκοσούρ το... θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ε, επιχείρημα ότι παραβιάζουν ε, τους κανόνες του ΠΟΕ. Όπως παραδείγματο χάρη τους παραβιάζει συστηματικά η Αργεντινή. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αργεντινή έχουν τεταμένες σχέσεις. Ε, ανησυχούμε ότι οδηγούμαστε σε διακρίσεις εναντίον των δικών μας επιχειρήσεων, του Ηνωμένου Βασιλείου δηλαδή, από την Αργεντινή. Δεν θα θέλουμε ε, να αφήσουμε τις αδικαιολόγητες οικονομικές δράσεις να συνεχίσουν έτσι. Ευχαριστώ. κύριος Ντάρντμοθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα επί ευκαιρία να αναφερθώ στη Βραζιλία. Ε, ε, το ΑΕΠ της είναι 48,3 εκατομμύρια δολάρια. Συγκριτικά το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχει ΑΕΠ 2,43 Τι ε, λένε τα μαθηματικά, οικονομία ε, του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το 97% της βραζιλιάνικης οικονομίας. Στο εμπόριο 37% των προϊόντων της Βραζιλίας είναι με άλλες χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής είναι πάρα πολύ αντίστοιχο και ε, συγκρίσιμο με το 40% του εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου με χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ Βραζιλία και Ηνωμένου Βασιλείου. Ουδή, απολύτω ουδή στη Βραζιλία θεωρεί ότι το 37% του εμπορίου της Βραζιλίας με υπόλοιπε χώρες Μερκοσούρ δικαιολογεί καθιοδήποτε τρόπο την ένταξη τη Βραζίλία σε μια πολιτική ένωση σε αντίθεση με αυτό, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επαγγελματίε πολιτικοί των κομμάτων του κατεστημένου ε, επανειλημμένα τονίζουν ε, ότι το 40% του εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου ε, που κατά τα άλλα μειώνεται ε, συνεχώς είναι από μόνο του ε, επαρκής δικαιολόγηση για να συμμετέχει η Βρετανία σε μια πολιτική ένωση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το επιχείρημα για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μόνο περίεργο, είναι κενό και τελείως έολο και ε, θα επανέλθω στο μέλλον σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε η ε, πρόθεση της πολιτικής ολοκλήρωσης στη Λατινική Αμερική ε, είναι εντυπωσιακή. Χειραφέτηση παγκόσμια σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα παρακολουθεί αυτά και να τα συνοδεύει θετικά. Στη Μερκοσούρ ε, επίσης υπάρχει μεγάλη σημασία και η ε, εταίροι μας, το τονίσατε, μας προσκάλεσε αυτή την ιστορική ε, διαδικασία να την συμπληρώσουμε και να την υποστηρίξουμε με μια σωστή συμφωνία των περιφερειών. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βραζιλία και άλλες χώρες Μερκοσούρ συμφώνησαν για εμπορικές συναλλαγές και οικονομική συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο και ε, αναζωγόνηση του γύρου της Δόχα. Όλα αυτά όμως τι απαιτούν. Να αναθεωρηθεί το ισχύον δόγμα ε, ότι θα πρέπει να προωθούνται μόνο τα εμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απέναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα τι απαιτεί. Από κοινού να ανταποκρινόμαστε στις κοινέ προκλήσεις. Δουλειά για όλους, παιδεία για όλους, έρευνα, επιστήμη, ανάπτυξη, καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, συνεργασία στο εμπόριο και στο περιβάλλον. Η ομάδα μου δεν μπορεί παρά να καταψηφίσει συμφωνίες που ενδιαφέρονται μόνο στην πρόσβαση των φυσικών πόρων ε, ορισμένων ολίγων. Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις της Αργεντινής και της Βραζιλίας μεταξύ άλλων δείχνουν ότι και εκεί όσο αυξάνεται η κρίση στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην ε, Ευρώπη υπάρχει ένα πολιτικό πνεύμα νέο που πνέει που θέλει να φέρει και πάλι την οικονομία στην υπηρεσία της κοινωνίας. Ευχαριστώ κυρία Ντότσου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μέχρι στιγμής ε, δεν ε, κατέληξαν σε αίσιο πέρα οι διαπραγματεύσεις και χαίρομαι για την ενημέρωση που μα έκανε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας είπατε κύριε Επίτροπε το πρωί ότι οι συνομιλίε αναμένεται να φτάσουν σε μια φάση που καλούμαστε να αποφασίσουμε αν θα ανταλλάξουμε προσφορέ ό,τι αφορά την πρέσβαση σε αγορέ αγαθών, υπηρεσιών και συμφωνιών δημοσίων προμηθειών. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ο πιθανό αντίκτυπο αυτή τη εμπορική συμφωνία για τη Βόρεια Ιρλανδία και άλλε χώρε που είναι εξαρτημένε από τη Γεωργία και ιδιαίτερα από τον τομέα βόλου κρέατο, ίσω ε, ε, πληγούν ολέθρια. Μία τέτοια συμφωνία θα κοστίσει στην Ευρωπαϊκή Γεωργία 30 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι βαρύτατο το τίμημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να μας ε, διαβεβαιώσετε και να μας καθησυχάσετε κύριε Επιτροπέ ότι δεν θα θυσιάσετε τη Γεωργία στο βωμό του, της εμπορικής συμφωνίας ε, όταν ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις για την, για την πρόσβαση στις αγορές. Είπατε στην αρχή ότι θέλετε μια ισορροπημένη, φιλόδοξη και περιεκτική συμφωνία με το Μερκοσούρ. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ε, μας και τους γεωργούς που εκπροσωπώ στη Βόρεια Ιρλανδία ότι σε αυτό το δεινό οικονομικό κλίμα ε, που αντιμετωπίζουν με αύξηση του κόστους ε, των εκμεταλλεύσεων και χαμηλά περιθώρια κέρδους και με πιθανή μείωση του γεωργικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη λίγη έμφαση που δίνουμε στην παραγωγή των τροφίμων. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υψώσει το παράστημά της προκειμένου να προσπίσει τα συμφέροντα των, συμφερόντων, τα συμφέροντα γεωργών στη Βόρεια Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ οι υπόλοιποι ομιλητέ και πρώτος ο κύριος Κρίστοφελ Φιέλναρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει θέση υπέρ των διαπραγματεύσεων. Είναι ένα πολύ επίμαχο θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά αν ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με το Μερκοσούρ, θα κερδίσουμε πολλά. Μιλάμε για 800 εκατομμύρια ε, καταναλωτές ε, συνδυαστικά Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει προστατευτισμός ακόμα στην τη Λατινική Αμερική. Ε, υπάρχει βέβαια και προστατευτισμό στην Ευρώπη, αλλά κυρίω στη Γεωργία, όχι αλλού. Ενώ εκεί γενικά υπάρχει ένα προστατευτισμό και, στα... και στη βιομηχανία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικέ λοιπόν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Ε, η περιοχή του Μερκοσούρ είναι πολύ σύνθετη περιοχή. Ε, για μας είναι προορισμός ε, γεωργικών προϊόντων μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά με αυτή τη συμφωνία, με χαμηλότερες ε, τιμές ε, γεωργικών προϊόντων για τους καταναλωτές μας και οι πολίτες του Μερκοσούρ μπορούν να έχουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες ε, τα οποία τα χρειάζονται σε πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι τώρα. Το θέμα είναι ότι οι διαπραγματεύσεις φέρνουν μεγαλύτερα μεγαλύτερε δυνατότητε για κέρδο. Αλλά αυτέ ακριβώ οι διαπραγματεύσει είναι πιο δύσκολε να τελεσφορήσουν. Εγώ σα καλώ, Επιτροπή, να μην κατεβάσετε τα χέρια και να έχετε και ένα σχέδιο καταφυγή, ένα σχέδιο Β. Ε, και στην Ασία κάποτε όταν διαπραγματευόμασταν είχαμε δυσκολίες. Είναι δύσκολο να διαπραγματευόμαστε γενικά με μια ολόκληρη περιοχή. Ίσως λοιπόν θα πρέπει λίγο τα πράγματα να τα δούμε μεμονωμένα. Ας δούμε ας πούμε τι γίνεται με την ε, Βραζιλία και ας εστιάσουμε καταρχήν εκεί. Ας εστιάσουμε σε κάποιους ε, τομείς, σε κάποιες χώρες. Ίσως θα πρέπει να συνεχίσετε λοιπόν αυτέ τι σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά να έχετε και ένα σχέδιο αναδίπλωση, ούτω ώστε να μην κολλήσουμε σε ένα θέμα και να σημειώσουμε γενική αποτυχία. Ευχαριστώ κύριο Λάγκε. Α, τώρα άναψε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για μένα η συζήτηση αυτή έχει τρεις λόγους να τη συζητήσουμε. Πρώτον, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι μάλιστα θέλουμε συνεργασία με τις χώρες Μερκοσούρ, διότι έχουμε πολλές κοινέ αξίες. Ο κύριος Σόλτς μίλησε για τα κοινά στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, ιδιαίτερα αυτό που κάνει η κυβέρνηση της Βραζιλίας. Έχουμε πολλά κοινά, έχουμε πολλές κοινέ οικονομικές υποθέσεις. Θέλουμε λοιπόν στενή οικονομική συνεργασία και εμπορική. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο μήνυμα της συζήτησης. Δεύτερον, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι χρειάζεται να ε, αποφασίσουμε και να διαλέξουμε πώς θα είναι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Πρώτον, να σκεφτούμε πάρα πολύ συγκεκριμένα ποιες χώρες ε, θα μπουν σε αυτό το καλάθι που διαπραγματεύεται η Ένωση. Και η Βολιβία θα μπει και ο Ισημερινός. Οι άλλες χώρες αυτό θα πρέπει γρήγορα να ξεκαθαριστεί για να ξέρουμε ποιος είναι ο συνομιλητής. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ε, σε αυτό το καλάθι. Δεν επιτρέπεται οι αξιώσεις και απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ε, συνάδουν και να απέχουν τόσο πολύ από αυτά που μπορούν να επιτύχουν και να ε, ε, φέρουν ως αποτέλεσμα οι χώρες Λατινικής Αμερικής. Και τρίτον, θα πρέπει να περάσουμε και στο διατάφτα. Ναι ή όχι. Δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευσης να διανοίζεται άλλη μια δεκαετία. Αυτά και σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ. Äh, im αυτή τη στιγμή ο κύριος Βλάσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ρητά και κατηγορηματικά ότι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων με το Μερκοσούρ είναι πολύ αργή και τα αποτελέσματα ισχνά και δυστυχώς ε, ούτε οι προοπτικέ είναι ιδιαίτερα ευίωνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ μια φιλόδοξη εμπορική συμφωνία με το Mercosur, βράχει πρόθεσμα. Επίση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην ε, απόρριψη των μέτρων προστατευτισμού. Γιατί η Αργεντινή και η Βραζιλία εφαρμόζουν τέτοια προστατευτικά μέτρα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην πετρελόβιομηχανία. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία. Να βρούμε συμμάχους στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου για να καταπολεμήσουμε αυτά τα αρνητικά μηνύματα του προστατευτισμού. Επίσης, να επικεντρωθούμε και στο θέμα της Βενεζουέλας και η νέα, η συμμετοχή, η νέα συμμετοχή αυτής της χώρας ε, θα περιπλέξει τα πράγματα. Ε, από τη στιγμή που θα ενταχθεί η χώρα αυτή θα πρέπει να δεχτεί τα συμφωνημένα ε, γιατί έχουμε συμφέροντα και εκεί. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε λοιπόν τι διαπραγματεύσει μα στα νέα οικονομικά συμφέροντα και τις νέες εξέλιξεις. Ευχαριστώ κύριος Όλτριχ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ε, του Μερκοσούρ συμμετέχουν σε μια τελωνιακή ένωση και είναι σημαντικό εμπορικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ε, ήδη ε, η Βραζιλία πριν από μερικά χρόνια είχε ε, εκδηλώσει το ενδιαφέρον για εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτελματωθεί από το 2010 και οι εξελίξεις είναι πολύ αργέ. Στι σημερινέ μα συζητήσει, θα πρέπει να αναλύσουμε τη βούλησή μας για προώθηση των διαπραγματεύσεων αυτό. Ε, επίκειται και η διάσκεψη κορυφής της επόμενης εβδομάδας στο Σεντιάγο της Χιλής. Ίσως ε, το περιεχόμενό της επηρεαστεί από τη σημερινή συζήτηση. Εκπροσωπούμε 500 ε, εκατομμύρια πολίτες και η Μερκοσούρ πολύ περισσότερους καταναλωτές. Σίγουρα αν οι εμπορικές μας συνδιαλλαγές ενταθούν, ίσως μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε από την οικονομική ύφεση. Θα πρέπει όμω οι χώρε του Μερκοσούρ να ανοίξουν τι αγορέ του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να επιλέξουν τελικά μια αρθολογική και ρεαλιστική συμπεριφορά προκειμένου να ευοδοθούν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα. Ο κύριος Φερέιρα. Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Το εμπόριο μπορεί να είναι ένα όργανο στήριξη τη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όμω, όταν δεν είναι ρυθμισμένο το εμπόριο, μπορεί ταυτόχρονα να καταστρέψει το εμπόριο, να οδηγήσει σε ύφεση και σε περιβαλλοντικέ καταστροφέ. Το άνοιγμα της μεγάλης αγοράς σε Μερκοσούρ ε, ενέχει κάποιες ε, αμφισημίες ε, και οι μεγάλοι οικονομικοί ομιλοί το γνωρίζουν και ποτέ δεν τα έχουν αρνηθεί είτε πρόκειται για το εθνικό είτε για το θεσμικό επίπεδο. Πρόκειται για τον προστατευτισμό κάποιων χωρών αυτής της περιοχής διότι υπάρχουν κυβερνήσεις και στη Λατινική Αμερική που υπεραμείνονται τις κυριαρχίες αλλά όχι των συμφερόντων των πολίτων. Αυτές οι χώρες τώρα διορθώνουν τις νέο φιλελεύθερες πολιτικές που τις οδήγησαν σε ύφεση και περιβαλλοντική καταστροφή. Τις ίδιες πολιτικές που εφαρμόζονται και στην Ευρώπη με τα γνωστά αποτελέσματα. Προσπαθούν να υπερασπιστούν λοιπόν, λοιπόν τα δικά τους τα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των πολιτών και γι' αυτό δεν υπάρχει καμία δυνατή συνενετική λύση. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Μπρόν. Uh, Παρότι δεν είμαι ενθουσιώδης οπαδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμα πρέπει να την έχουμε, καλύτερα να είναι κανείς περισσότερο Ευρωπαίος παρά λιγότερος. Αυτές οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ και διαφόρων άλλων εμπορικών ενώσεων δεν εστιάζονται αποκλειστικά στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρώπη. Έχουν μια παγκόσμια πτυχή, όλοι οι κοσμοπολίτες νέοφιλελεύθεροι δεν γνωρίζουν καμία διαφορά ανεξαρτήτως ο χώρας και επιθυμούν να κυκλοφορούν οι άνθρωποι και οι υπηρεσίε χωρί κανένα πρόσκομα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα ότι οι λαοί και διαφορετικέ παραδόσει θα εκλείψουν και τα πρότυπα ζωή θα εξισωθούν προ τα κάτω σε ένα επίπεδο που δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο ζωή των Ευρωπαίων. Ολόκληρο ο κόσμο θα είναι πλουσιότερο αλλά για του ισχυρότερου και σίγουρα αυτό δεν ισχύει για μεμονωμένε χώρε ή συγκεκριμένε κοινωνικές ομάδες ε, και τομείς που επίσης ε, δεν θα είναι πλουσιότεροι. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ένωση Μερκοσούρ δημιουργήθηκε το 1991. η εντολή που έχουμε εμείς προέρχεται από του ε, υπουργού των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέρχεται στο 1999. Νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να επικυρώσουμε και πάλι αυτή την εντολή από το Συμβούλιο των Υπουργών, γιατί από το 1999 οι οικονομικέ συνθήκε έχουν αλλάξει. 12 πρόσθετα κράτη-μέλη έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα που μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αρμοδιότητα και στι εμπορικέ συμφωνίε. Λυπάμαι για την απουσία του Συμβουλίου, το οποίο θα έπρεπε να είναι παρόν σε αυτή τη συζήτηση επί τη ουσία. Η εντύπωση που έχω είναι ότι τα δύο αυτά εμπορικά μπλοκ κινούνται προς μια αμοιβαία καχυποψία. Το μπλοκ των χωρών Μερκοσούρ έχει λιγότερη εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της χρηματοδημοσιονομικο-νομισματικής αναταραχής που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Βλέπετε ότι η πρόοδος της Βασιλείας λέει σε όλα τα διεθνή φόρα ότι είναι η δική της η Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική που, αναβαθμί, οδηγεί σε ανατίμηση του ΡΕΑΟ. Θα πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έχουμε πραγματικούς λόγους να είμαστε καχύποπτοι, γιατί έχουν ε, αναστείλει την παρουσία της Παραγουάης με τρόπο ο οποίος θα είναι παράνομος, χωρίς να πούν τίποτα. Η προσχώρηση της Βενεζουέλας μπήκε παράνομα, χωρίς να πούνε τίποτα. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αλλαγές που έχουν επιφέρει στη συμφωνία έχουν επιφέρει προστατευτισμό. Επίσης και για τις νήσους Μαλουίνες, Παύλα, Φάλκλαντ, υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να μπορέσει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να μπορέσει να είναι στη βάση μια συμφωνίας ε, σύνδεσης, η οποία να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γιάννη ε, Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω την ε, ιστορική αυτή συμφωνία η οποία θα συναυθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ε, με την Λατινική Αμερική μέσω της Μερκοσούρ. Το να συμφωνήσουν 800 εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτεί να ληφθούν πολλά πράγματα υπόψη, δεδομένου ότι το θέμα του εμπορίου δεν είναι εύκολο. Το είπαν όμως δύο γυναίκες το 2010. Η Μαρία Τερέζα Φερνάνδες Δελαβέγκα, η αντιπρόεδρο ε, τη Ισπανία, και πήγε στην Λατινική Αμερική, συμφώνησε με την Κριστίνα Φερνάντε και έτσι ξαναξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει. Ελπίζω λοιπόν τώρα στη Χιλή οι γυναίκε κυρίω όπου είναι πάρα πολύ πρακτικέ, η κυρία Μέρκελ, η κυρία Ρούσελ, η είπατη Εκπρόσωπο, ε, η πρόεδρο Αργεντινή, να αναζητήσουν έναν τρόπο προκειμένου να ε, ξεμπλοκαριστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να φτάσουν σε αίσιο τέλος. Διότι το πρόσκομα δεν είναι τεχνικής φύσεως, δεν είναι διαδικαστικής φύσεως. Κατά την άποψή μου δεν είναι τη μιας ή της άλλης χώρας, είναι απλώς έλλειψη πολιτικής βούλησης στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ίδιοι οι διαπραγματευτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση μα τολούν, διότι εγώ προεδρεύω στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα με τη Μερκοσούρ και μα λένε ότι χρειάζεται να ξεπλοκαριστούν τα πράγματα Προ τα πάνω από τους πολιτικούς, από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ελπίζω λοιπόν κύριε Επίτροπε και είμαι βέβαιο ότι και εσείς το ίδιο ελπίζετε ότι στη Χιλή θα ε, σταματήσει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριος Aylward. Χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία να τονίσω και πάλι την αντίθεσή μου στην συμφωνία αυτή. Η εμπειρία μας από το παρελθόν είναι αρνητική. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν επιμένει στο να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Είπε η Κομισιόν ότι ο τομέας της μεταποίησης θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Θα έχει θετικά αποτελέσματα, αλλά τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τη στιγμή αυτή δείχνουν <clears throat> ότι θα υπάρξει μεγάλη επίπτωση στον αγροτικό τομέα που θα οδηγήσει σε απόλυτες θέσεων απασχόλησης. Υπάρχουν σημαντικές απώλειες στον τομέα του βοήου κρέατος και επιπτώσεις στις άλλες αγροτικές παραγωγές. Η γεωργία είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της αγροτικής ζωής και του αγροτικού τρόπου ζωής και πρέπει να προασπιστεί. Όλοι αυτοί που υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα θεωρούμε ότι είμαστε προστατευτιστές, αλλά η αγροτική οικονομία είναι η ραχοκοκαλιά οικονομιών όπως η Ιρλανδία και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η βάση για το μέλλον μας. Δεν μπορούμε λοιπόν τα επόμενα χρόνια, όταν προβλέπεται και αύξηση του πληθυσμού τη γη, να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δημογραφική αύξηση χωρί τη σωστή αγροτική ε, δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, παροτρύνω του ηγέτε Ευρωπαϊκή Ένωση και εσά, κύριε Επίτροπε, να μην θυσιάσετε στο βωμό των συμφωνιών αυτών την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν εν ζωή η γεωργή και η γεωργική δραστηριότητα. Ευχαριστώ, κύριο Νίκολσον. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το θέμα αυτό μπορεί να οδηγήσει στο άνοιγμα του κοιτίου της Πανδώρας σε σχέση με τα αγροτικά θέματα και την ε, οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω αυτά τα πράγματα. Πριν από λίγα χρόνια πήγα στη Βραζιλία και είδα με τα δικά μου τα μάτια αλλά πέ, ότι αντίθετα από αυτά που μας λέει η Κομισιόν και μας διαβεβαιώνει για όλα αυτά ότι η Βραζιλία είναι το τέλειο μέρος για την παραγωγή βοήου κρέατος είναι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, τα θέματα ανιχνευσιμότητας που αφορούν και τη Βραζιλία και την Αργεντινή δεν έχουν ε, τα ίδια πρότυπα όπως στην Ευρώπη. Πολλές φορές είναι καλύτερα κιόλα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα προκύψουν για το τομέα του βοήου κρέατος. Εγώ δεν θα αλλάξω άποψη για τα θέματα αυτά για χώρες όπως είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή σίγουρα δεν ισχύουν τα ίδια πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προϊόντα αυτά λοιπόν δεν θα πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια θέση αρχής και δεν θα πρέπει ποτέ να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Αγκουράκης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσει στη Μερκοσούρ ώστε να αποδειχτεί επιτέλου τη σύναψη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Πρόκειται για την οικονομική πολιτική πλευρά τη υπεριαλιστική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αλλού ασκείται με την ομή στρατιωτική βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάμψει τι λαϊκέ αντιστάσει, γιατί οι συμφωνίε επιβάλλουν ιδιωτικοποίηση, αρπαγή πρώτων υλών και αγορών για τα βιομηχανικά προϊόντα και τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρο των ντόπιων συνοδεύεται από λαιλασία της παραγωγικής βάσης ένταση της εκμετάλλευσης καταστροφή των φτωχών αγροτών των εργατών γης και των αυτόχθονων πληθυσμών. προκαλεί πληγές στο περιβάλλον. η πλειοψηφία του ευρωκοινοβουλίου με το κοινό ψήφισμα στηρίζει τις επιδιώξεις των μονοπωλίων της ευρωπαϊκής ένωσης για έξοδο από την καπιταλιστική κρίση στις πλάτες των λαών αυτή η πολιτική όμως είναι και επικίνδυνη. το λέω αυτό γιατί προωθεί την αντιπαράθεση μεταξύ των χωρών της περιοχής την υπονόμευση της ελάκ των κυβερνήσεων της κούβας και της βενεζουέλας που αντιστέκονται στους σχεδιασμούς αυτούς. ταυτόχρονα οξύνει τους ανταγωνισμούς με τη ΣΥΠΑ και τις χώρες της ομάδας brics. ομάδα του ΕΛΚ Η κυρία Κέστιγκερ, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αυτή η συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ και προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτή τη συμφωνία με στην νέα της μορφή. Αλλά έχουν και πάλι τελματωθεί οι διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να υπάρχει αμοιβαιότητα στις συμφωνίες οι οποίες, οι οποίες συνάπτονται και όταν πρόκειται για εμπορικού εταίρου που έχουν μεγάλη εμπορική σημασία και οικονομική σημασία. Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν δεν υπάρχει το αντίβαρο για αυτή την συμφωνία. Οι μελέτε και τη Κομισιόν τη ίδια καταδεικνύουν ότι θα υπάρξει μεν μία ένα κέρδος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλά υπερκεράζεται από την απώλεια στον αγροτικό τομέα που υπολογίζεται σε 7 δισεκατομμύρια. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη της λοιπόν η Κομισιόν και το έχουν τονίσει και διάφοροι συνάδελφοι ότι δεν μπορεί να θυσιαστεί ο αγροτικός τομέας με τέτοιες συμφωνίες. Γι' αυτό επαναλαμβάνω την, ε, την πρότασή μου ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν ρήτρε διασφάλιση σε όλα τα κεφάλαια που αφορούν τι ε, αγροτικέ συμφωνίε, ώστε στι παραγωγέ τρίτων χωρών να ισχύουν τα ίδια πρότυπα κοινωνικά και περιβαλλοντικά όπω ισχύουν και για τα αγροτικά ε, θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να σα ρωτήσω, κύριε ε, Επίτροπε, θα λάβετε υπόψη την έννοια τη βιωσιμότητα και τη αηφορία στι διαπραγματεύσει για τα αγροτικά θέματα, όπω έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του. Και επίσης υπάρχει και κάποιο εναλλακτικό σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των ε, εντάσσεων που παρατηρούνται στις χώρες της Μερκοσούρ για μεμονωμένες συμφωνίε με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κούτας. Ευχαριστώ. Ε, η Μερκοσούρη είναι ο 8ος εμπορικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυξηθεί οι εμπορικές συναλλαγές τα περασμένα χρόνια. Ε, και πέρσι αναδείχθηκε στο πρώτο εμπορικό εταίρο και πρώτο επενδυτή στην περιοχή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση με αυτόν τον τρόπο και θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για τη σύναψη εμπορική συμφωνία. Νομίζω ότι είναι θετικό και για τι δύο περιοχέ αυτού του κόσμου. Λοιπόν, η έναρξη και πάλι των διαπραγματεύσεων, ε, η ολοκλήρωση μάλλον των διαπραγματεύσεων ε, το 2010 και τη δημιουργία οικονομικού χώρου ήταν θετικό βήμα, όμω εξακολουθούν να υπάρχουν προστατευτικά μέτρα σε διάφορου χώρε τη περιοχή. Στο Σαντιάγκο τη Χιλή την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω, Επίτροπη, στις διαπραγματεύσεις που θα συμμετάσχετε να επικρατήσει η βούληση διαλόγου και εξέβρεση μιας συμβαστική λύσης. Ευχαριστούμε κύριος Δίας Δεμέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μάιο συμπληρώνονται τρία χρόνια από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην πραγματικότητα. Εγώ προσυπογράφω απόλυτα την ε, επιτυχή τους κατάληξη. Θα ήθελα όμως να σας πω τα εξή, κύριε Πρόεδρε. Η περιοχή της Μερκοσόρ είναι η περιοχή που παράγει περισσότερα προϊόντα με τον κόσμο και υπάρχουν και τα περισσότερα ενεργειακά αποθέματα παγκοσμίω. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα και η σημασία αυτής της διαπραγμάτευσης ε, μεταξύ των εταίρων. Το φθινόπωρο μεταβήκαμε στη Βραζιλία και εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μεν μια θετική στάση αλλά ταυτόχρονα και μια αμφίσιμη στάση. Ο κύριος Επίτροπος μας είπε ε, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τι πρόοδος έχει υπάρξει στα πλαίσια της νομοθεσίας, αλλά αυτό στην Ισπανία είναι ουσιαστικά το να θολώνουμε τα νερά. Το θέμα είναι κατά πόσον θα προχωρήσουμε τα βιομηχανικά και γεωργικά ζητήματα και αν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα συμφέροντά μα και αν θα προχωρήσουμε και στο θέμα των υπηρεσιών. Αυτό που σα ζητώ λοιπόν κύριε Επίτροπε και είναι η τρίτη φορά που αναφέρεται το θέμα τη πολιτική βούληση εδώ στην Ολομέλεια σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν στη Χιλή να επιδείξετε κι εσείς ε, την πολιτική βούληση και να βοηθήσετε και του υπολείπους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είμαστε και εμείς στο Σαντιάγο της Κυλή και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και στη συνέχεια θα ήθελα να έρθετε εδώ στην Ολομέλη για να μπορέσουμε να γνωρίζοντας ε, να αποφασίσουμε. Να αποφασίσουμε αν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ή αν θα ακολουθήσουμε την εναλλακτική λύση, να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να συνάψουμε διμερεί συμφωνίες. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μεσή, ο κύριος Μίρσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεγκούχτ, ελπίζω ότι ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων υπήρξαν δυσκολίες. Έχετε προετοιμάσει κάποιες συμβιβαστικέ προτάσεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει προετοιμαστεί πλήρως το θέμα αυτό των συμφωνιών με τη Μερκοσούρα από την πλευρά της Κομισιόν. Γι' αυτό έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι ικανοποιητική. Θυμηθείτε ότι έχουν υπάρξει ε, δράσεις αντι-dumping από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της Ινδονησίας αλλά και της Αργεντινής. Χρειαζόμαστε πιο επαγγελματικού χαρακτήρα με την χιλή. Αν δεν μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Μερκοσού, τότε θα πρέπει να αλλάξετε ομάδα διαπραγματευτών. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάγκλα έχει το λόγο. <coughs> κύριε Πρόεδρε. Και ιδίω μετά από την συμφωνία μας με την Κολομβία, το Περού και την Κεντρική Αμερική, θα πρέπει να προσέξουμε ότι η σχέση μας με την πιο σημαντική εμπορική δύναμη της περιοχής, τη Μερκοσούρ, να είναι πάντα στο κέντρο της προσοχής μας. Πρέπει να τηρηθούν βασικές δημοκρατικές αρχές όπως είναι τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα του περιβάλλοντος βέβαια. Η Μερκοσούρ μαζί με την ε, ε, Βραζιλία, μια από τις χώρες BRIC, είναι από τους πιο ισχυρούς οικονομικούς πόλους του κόσμου. Αυτό δίνει μια τεράστια δυνατότητα και δυναμικό ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των εμπορικών της σχέσεων και επίσης δίνει δυνατότητα καλύτερων οικονομικών και πολιτικών σχέσεων. Αυτό όμως θα μπορέσει να οδηγήσει σε κάποια κέρδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση άμα τηρηθούν ορισμένοι βασικοί κανόνες ο βασικό κανόνα για τι εξωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι οι δημοκρατικέ αρχέ, του κράτο δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ οι προδιαγραφέ σε επίπεδο περιβάλλοντο και εργασιακών θεμάτων. <clears throat> Είναι πολύ σημαντικά τα προϊόντα στο γεωργικό τομέα της Νότιας Αμερικής, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν μέσα στα πρότυπα των ευρωπαϊκών ε, προτύπων για τη γεωργική παραγωγή για να είναι αποδεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί υποστηρίζουμε τη συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Μερκοσούρ αν τηρηθούν όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και αν <clears throat> και οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές είναι διαθέσιμοι να προχωρήσουν σε μόνιμο τρόπο προς μια προσέγγιση στα θέματα αυτά. Ο κύριος Κάπολο Σάντους έχει το λόγο. Το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχίζοντας ε, να συγχαρώ τον κύριο Μωρέιρα, τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΙΝΤΑ, για την αρχική παρέμβασή του σε αυτή τη συζήτηση. Συμφωνώ απολύτως. Θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε για την επιτακτική ανάγκη να προωθήσουμε μια μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση ανάμεσα στα διάφορα οικονομικά μπλοκ σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, εξασφαλίζοντας έτσι ειρήνη και ευημερία σε διεθνή κλίμακα. Πάντω στην περίπτωση του Mercosur οι δυναμικέ που έχουν δημιουργηθεί έχουν θετικό αποτέλεσμα σε κάποιου τομεί. σε άλλου πάλι ξεκάθαρα έχουν αρνητικά αποτελέσματα και κυρίω λείπει ένα θετικό αποτέλεσμα για του πολίτε, για την αξιοπρεπή ζωή του και τα πρότυπα ζωή του. Ε, το ίδιο θέμα αντιμετωπίζουμε και στον τομέα τη Γεωργίας Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα τη αγροβιομηχανία θα πρέπει να καρποφορήσουν αυτέ οι προσπάθειε. Ε, αυτό σίγουρα δεν ισχύει για τους γεωργούς ε, που παράγουν την πρώτη ύλη κυρίως σε συγκεκριμένου ε, τομεί, όπως το λάδι και το ξύδι. Ε, για το στον τομέα της βιομηχανίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα μελετήσει το ψήφισμα που κατά πάσα πιθανότητα θα υπερψηφιστεί με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Χαιρόμαστε διότι καλύπτει όλες τις ανησυχίες που έχουμε και τις προσδοκίες που έχουμε για τις θετικές επιπτώσεις της συμφωνίας με το Mercosur. Σας ευχαριστούμε. Ζάλμπα Μπίντεγκάιν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρώπη έχει έναν φυσικό εμπορικό σύμμαχο στην Αμερικανική Υπέρο λόγω πολιτισμού, γλώσσας και λόγω άλλων δεσμών τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση και μια συνέχεια των σχέσεών μας. Η Μερκοσούρ είναι το τέταρτο πιο σημαντικό οικονομικό μπλοκ ε, παγκοσμίω. Είναι το 80% του ΑΕΠ της ε, περιοχής και έχει πάνω από 40 εκατομμύρια κατοίκου. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το 2010 ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να ε, υπερβούμε τα προσκόμματα προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας ε, που είναι μια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας και να υπάρξουν αμοιβαία ωφέλη. Στη διαδικασία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι εμπλέκεται πολύ στενά και θέλει να προχωρήσει με ε, συνδυασμένο τρόπο για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα από τα ε, θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα είναι οι επενδύσεις. Οι άμεσες επενδύσεις στη Μερκοσούρ είναι περισσότερες αθρηστικά από τις επενδύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα ή στη Ρωσία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε μέσω προστασίας αυτών των επενδύσεων. Να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική αλληλεξάρτηση και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Γι' αυτό ακριβώς και χρειάζεται, όπως ακούστηκε εδώ σήμερα, να υπάρχει πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι προς όφελος όλων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κύριος Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, Δεδομένων των πολυέρευμων και συνεχών διαπραγματεύσεων που γίνονται χωρίς ε, να έχουμε κανένα αποτέλεσμα τα τελευταία δύο χρόνια, καταλαβαίνετε πόσο έντονη είναι αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ για τα γεωργικά προϊόντα. Αφενός η Μερκοσούρ πιέζει για να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης των γεωργικών της προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ίσως ε, να έχει εμπορικές διευκολύνσεις για τα μεταποιημένα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα διπλωματικό μπραντεφέρ όπου για πολλωστή φορά και πάλι ε, κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι Γεωργοί οι οποίοι είναι στο έρμεο αποφάσεων και διαπραγματεύσεων που ε, εξαρτώνται από άλλους τομείς. Πρόκειται για ένα τομέα λοιπόν ο οποίος ε, τιμωρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ εμείς με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική ε, προσπαθούμε να τον έχουμε σε υψηλή προτεραιότητα ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε στους πολίτες υγιή και ανοιχνεύσιμα προϊόντα και στους γεωργούς κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην υποκύψουν στην ανταγωνιστικότητα των ε, ε, γεωργικών προϊόντων στις ε, ευρωπαϊκές αγορές. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις, στις υπόλοιπες διμερείς συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην θυσιάσουμε την ε, ε, ευρωπαϊκή γεωργία στο βωμό μιας έντονης προσπάθειας, όπως μου φαίνεται ότι γίνεται σε αυτή την περίπτωση στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Ευχαριστώ κύριος Καντά, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είναι προφανές ότι έχουμε δύο μεγάλα οικονομικά μπλοκ όπως είναι η Ευρώπη και η Μερκοσούρ, ότι έχουν συμφέρον να έχουν ισχυρές σχέσεις εταιρικού χαρακτήρα και είναι προς το συμφέρον μας να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά όπως ελέγχθη ήδη από πολλού συναδέλφου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα <clears throat> στην εξέλιξη της Ευρώπης αφενό και της ε, Λατινικής Αμερικής από τη στιγμή που εδόθη η αρχική εντολή. Δεν έχουμε την ίδια οικονομία, δεν έχουμε τους ίδιους ανθρώπους και είναι απαραίτητο, όπως τονίστηκε από πολλούς, να υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση της εντολής. Πρέπει μέσα στο νέο πλαίσιο να υπάρχουν εγγυήσει για τα μέτρα αμοιβαιότητα τα οποία θέλουμε να υπάρχουν και από τι δύο πλευρά για την προστασία των καταναλωτών. Είδαμε του τελευταίου μήνε ότι οι χώρε τη Νότια Αμερική δεν έχουν δεν ντρέπονται καθόλου να εφαρμόσουν προστατευτικά μέτρα όταν αυτό τους βολεύει. Εμείς Θέλουμε όχι μέτρα προστατευτικά, αλλά μέτρα τα οποία θα προστατεύουν την υγεία των καταναλωτών στον υγειονομικό τομέα. Ξέρουν ότι οι καταναλωτέ μα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουν. Ευχαριστώ, κύριο Γκλάτφελντερ. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα δεν έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσούρ. Έχουμε προσκρούσει σε ένα τείχο ουσιαστικά. Έχουμε πάρα πολλά εμπόδια σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που είναι, σφαλ, που είναι φταίξιμο της ίδιας Μερκοσούρ. Εθνικοποιούν ευρωπαϊκές εταιρείες, <clears throat> έχουν ε, διαμφισβητήσει την ε, ταφική ακαιρεότητα ορισμένων χωρών μέσα στη Μερκοσούρ και έχουν δεχθεί και την Βενεζουέλα στους κόλπους τους. Η αρχική διαπραγματευτική εντολή ήδη δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής. Πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με χώρες με τις οποίες έχουμε κάποια ελπίδα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συνταχθεί μια νέα διαπραγματευτική εντολή, η οποία λαμβάνει υπόψη τις ε, ευαισθησίες των γεωργών μας και των αγροτικών μας προϊόντων, τα θέματα της ε, ασφάλειας των τροφίμων και της ευζοίας των ζώων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την τωρινή Κυρία Ραφ Γκαρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μερκοσούρ θα πρέπει να θεμελιώσουν και να προωθήσουν τις διμερείς τους σχέσεις και ε, οι δύο έχουν συμφέρον να προχωρήσουν τις εμπορικές σχέσεις. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι οι συνέπειες ε, του να ανοίξει περισσότερο κοινοτική αγορά σε γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τις χώρες αυτές. Ιδίω ε, στα θέματα του βόηου ε, κρέατος ε, στα πουλερικά στα όσα συζητήσαμε στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων ε, δεν έκρυβα τις επιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε στις αναφορές που έκαναν οι χώρες της Μερκοσούρ στο γεωργικό τομέα. Ε, σύμφωνα με τα διάφορα κράτη-μέλη μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική πτώση αλλά ε, υπολογίζεται ότι θα χαθούν 33.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εισρωή των προϊόντων αυτών. Και να σας πω ότι ε, αυτά είναι πολύ πιο αισιόδοξα από τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε αγορές στον τομέα του βόλου κρέατος και των πουλερικών χωρίς να απαιτείται αμοιβαιότητα. Και οι συμφωνίες με τη Μερκοσόρ θα πρέπει να βασίζονται στην κοινή γεωργική πολιτική και στα όθια σας διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε στην διαδικασία ad hoc βάσει της οφθαλμοσυλληπτικής διαδικασίας. Η κυρία Πετράγνου ήδη έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην, στο να δοθεί νέα όθηση στην οικονομία, να παραχθεί πλούτος και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόληση. Η γεωργία επανειλημμένα χρησιμοποιείται ως ένα νόμισμα για ε, τις συναλλαγές ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία. Στι σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ βλέπουμε στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 τις ε, που θα υφίστατο μετά τη σύναψη της συμφωνίας η Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και απορρίφθηκε από τους γεωργούς διότι μειώνεται το εισόδημά τους και η ίδια τους η παραγωγή. Και πέραν αυτού η αγροβιομηχανία εποφελείται ε, από την ολοκλήρωση νέας αγοράς και το ίδιο και οι καταναλωτές ε, έχουν καλύτερη υγιεινή, καλύτερη ποιότητα στα τρόφιμα, προστατεύονται τα ζώα και το περιβάλλον. Ε, βέβαια σε ευαίσθητες περιοχές υπάρχουν μεγαλύτερη μεγαλύτερε ζημιέ ε, και το ίδιο ισχύει και για κάποια προϊόντα όπω το κρέα ε, στι Ασόρε. Ε, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με μία κρατεά γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επισητιστική ανεξαρτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεμελιώδε από πλευρά πολιτική. Αυτέ οι πτυχέ θα πρέπει να συνυπολογιστούν οπωσδήποτε εν ώψη σε ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Σα ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Λουίς ε, Πάολο Άλβες ε, τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αγνοήσει ή να μην υπολογίζει κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, του ψηφίσματος του Μαρτίου του 2011 για τη Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Εμπόριο που προτείνονται επίσης και στο ψήφισμα για το Μερκοσούρ, μάλλον που παραλείπονται τώρα στο ψήφισμα για το Μερκοσούρ. Στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε τη γεωργία για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς ε, αγορές. Ε, το εμπορικό έλλειμμα στα γεωργικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπερεύει πλέον τα 7 δις και δεν μπορούμε να σκάψουμε περισσότερο αυτό το χάσμα που υπάρχει και να υποσκάπτουμε έτσι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου. Έχουμε ήδη μελετήσει τις επιπτώσεις αυτής της Ευρωπαϊκής ε, Συμφωνίας ε, σε εδαφικό επίπεδο και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι σε περιοχές απομακρυσμένες ε, όπως οι Ασόρες υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστούμε κυρία Τσίκαου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούσε το 2009 ότι η Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας ε, για τις μεταφορές θα είχε 460.000 επιπλέον επιβάτες για ένα χρόνο και αντίστοιχα ωφέλη. Ε, και ότι η συμφωνία αυτή θα είχε και θετικές επιπτώσεις και θα είχαμε δημιουργία ε, θέσεων εργασίας. Εκτιμάται ότι θα έχουμε 9.800 νέες θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, ε, κύριο Επίτροπε ως ε, εισηγητρία για τα θέματα της Συμφωνίας για τις Αεροπορικές Μεταφορές τι περιμένετε να έχουμε ως αποτέλεσμα. στη τελευταία υπουργική διάσκεψη στο Μερκοσόρ που θα γίνει στα τέλη Ιανουαρίου σκοπεύετε να συζητήσετε και τη συγκεκριμένη συμφωνία προκειμένου να γίνει κάτι για τις διαπραγματεύσεις. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ θα πρέπει να επικεντρωθούν και σε κοινέ πρωτοβουλίες προκειμένου να αναπτυχθεί η παραγωγή και θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, μπορώ να ζητήσω από τον κύριο Επίτροπο να λάβει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν εκπλήσωμαι από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους έντιμους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Βλέπω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστηρίζει τις ε, διαπραγματεύσεις σε σοβαρό επίπεδο με τις χώρες Μερκοσούρ, αλλά το ταγκό χορεύεται από ζευγάρι. Πρέπει και οι δύο πλευρές να συμμετάσχουν. Και οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τις διαπραγματεύσεις είναι γνωστοί σε εσά. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει πολιτική θέληση, το πολιτικό περιθώριο, η χορευτική δυνότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε χάσει το παιχνίδι τελείως, δεν νομίζω. Γιατί οι Βραζιλιανοί έχουν προβεί σε μια νέα επισκόπηση της δραστηριότητας τους στα βιομηχανικά θέματα και οι βιομηχανικοί κύκλοι έχουν αντιμετωπίσει την συμφωνία αυτή πολύ πιο θετικά από ό,τι πριν από δύο ή τρία χρόνια. Δεν πηγαίνουν όλα προς την λάθος κατεύθυνση. Ίσως θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά όμως δεν ξέρω. Περιμένω λοιπόν τη συνάντηση στο Σαντιάγο της Χιλής για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο φως το οποίο θα ρηφθεί στα θέματα αυτά. σε σχέση με τα θέματα, με τα ερωτήματα τα οποία διατυπώθηκαν για τα αγροτικά θέματα. Δεν εκπλήσωμε για όλα αυτά. Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε τη Γεωργία. Το μόνο που λέω είναι ότι, ότι και σίγουρα δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσουμε ως κατά κάποιο τρόπο ανταλλακτικό εργαλείο τη Γεωργία. Αλλά οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ πολλών τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Η Γεωργία δεν είναι ο μόνος τομέας ο οποίος εμπίπτει σε αυτή τη συμφωνία, ένας νευραλγικός τομέας. Δεν μπορεί να κάνει όμως κανείς μια συμφωνία μόνο για τα βιομηχανικά προϊόντα ή μόνο για τα αγροτικά προϊόντα. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία για τα θέματα αυτά. Και φυσικά ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία σε όλες αυτές τις συμφωνίες και αυτό θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι η παγκόσμια αγορά για τα αγροτικά προϊόντα προχωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση και για πρώτη φορά <clears throat> οι αγροτικές μας εξαγωγές οδηγούν σε ένα πλεόνασμα. Ας είμαστε λιγάκι λιγότερο λοιπόν αμυντικοί στα θέματα αυτά και είναι υπερβολικές οι δηλώσεις για εκατομμύρια για χιλιάδες θέσεων εργασίας που θα χαθούν. Μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λογική συμφωνία με τις χώρες Μαρκοσούρ, εφόσον έχουν την πολιτική θέληση και την δυνατότητα να το πράξουν από τη δική τους πλευρά. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, θα το πράξουν. και δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτό το οποίο είπαν ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου, το εναλλακτικό σχέδιο, το σχέδιο ΒΟ, δεν έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο βου αυτή τη στιγμή. Και είναι πολλές χώρες στη ζώνη του Μερκοσού που ούτε και αυτές έχουν κάποια αναλλακτική δυνατότητα. Αυτά δεν τίθενται επιτάπητος αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ακόμα για συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μερκοσούρ ακόμα. Αλλά ο χρόνος τρέχει. και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ατερμόνως με τα θέματα αυτά. <clears throat> Θα πρέπει οι χώρες Μερκοσού να αποφασίσουν τι θέλουν, ποια είναι η θέλησή τους και ποιοι είναι οι στόχοι τους και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ αυτών των δύο πολύ σημαντικών εμπορικών ομίλων και οντοτήτων. Ας περιμένουμε λοιπόν τη συνάντηση επόμενης εβδομάδας στο Σαντιάγο και εγώ θα σας δώσω μια αναφορά όταν επιστρέψω στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Για το κλείσιμο αυτής της συζήτησης έχουν παρουσιαστεί τρία ψηφίσματα τα οποία θα ψηφιστούν στις 12 το μεσημέρι. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης και θα ήθελα να σας κάνω δύο ανακοινώσεις από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Μία ανακοίνωση αφορά την αίτηση των Ολλανδικών Αρχών για την άρση της ασυλίας του κ. Κράτσμαν βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6 παράγραφος 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραπευθεί αυτή η αίτηση στην Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δεύτερη ανακοίνωση